σας ε, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι. Ξεκινούμε λοιπόν αυτή την μακρά συνεδρία ψηφοφοριών. Γραπτή δήλωση των Μπεσέ, Ντερί, Κάινεμ και Οκτάβια Σάρδο σχετικά με την ε, μεταχείριση των παραγών ε, ορνήθων. Έχουν ήδη, έχει ήδη υπερψηφιστεί από την πλειοψηφία και βάσει του άρθρου 122 του κανονισμού ε, θα μεταδοθεί αρμοδίως με την ένδειξη όλων των ονομάτων που έχουν προσυπογράψει στα πρακτικά. Έχουμε τώρα την, ε, ε, την Σενίσκη Μπεζέ Όνιμπολ Τάκουλα σχετικά με μεγαλύτερη ε, στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για, τα, ε, για τον αθλητισμό. Και βάσει του άρθρου 123 και το θέμα αυτό θα δημοσιευθεί στα πρακτικά της επόμενης συνεδρίας. Ο κύριος Κέλλη μπορεί να μιλήσει για 30 δευτερόλεπτα. Παρακαλώ κύριε Κέλλη. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε εξ ονόματος όλων των υπογραφόντων του Ιβο Μπαλέτου Χανού Τάκουλα, της Μαρίας Χάνεμπολ και άλλων θέλω να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που υπέγραψαν αυτή τη δήλωση. Είναι σημαντικό ότι περίπου 50% αυτών που υπέγραψαν ήταν γυναίκες. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν πάρα πολύ όλους αυτούς που συνεργάστηκαν σε αυτό το εγχείρημα και να αποτίσω ιδιαίτερο <clears throat> φόρο τιμής σε αυτούς οι οποίοι έπαιξαν ρόλο σημαντικό σε, στην ε, υπογραφή αυτού του ψηφίσματος. Ευχαριστώ πολύ. Γραπτή δήλωση 61 του 2010 υποβληθήσα από τους συναδέλφους Τόμσεν, Λίνε, Φεγγερέιδο, Ντέλη και πρώτα ο κύριος Ντέλη έχει ζητήσει το λόγο. Πρόκειται για την στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους αστέγους. Ε, σύμφωνα με τον κανονισμό 123 ε, θα μεταδοθεί και θα δημοσιευθεί στα κείμενα της ε, προηγούμενης Ολομέλειας. Για 30 λεπτά Καρίμα Ντελή. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, με μεγάλη συγκίνηση εξ ονόματος των συναδέλφων Τόμσεν, Λίνεφ, Γκυρέιδο και Πρότασιεβίτσε θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την στήριξη ε, που δώσατε στην δήλωση 61-2010. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, στην ε, ε, εμβληματική της πρωτοβουλία παρουσιάζει μια πλατφόρμα για τους άστεγους. Νομίζω ότι έφτασε η ώρα να ξεχάσουμε τα ωραία λόγια. Πρέπει να περάσουμε στις πράξεις. Συγκεκριμένες προτάσεις θα πρέπει να εφαρμοστούν έτσι ώστε το 2015 κανένας άστεγος πια να μην κοιμάται στους δρόμους. Καλά Χριστούγεννα, ευτυχισμένες γιορτές και σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Έχει ζητήσει το λόγο ε, ο κύριος Μπεσέ. Ε, Εξ ονόματος των τριών συναδέλφους ε, μου Πετικάνεν, ε, Σαρμπού και Ντέιβις θα ήθελα να ευχαριστήσω τους 410 βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ε, ε, υπέγραψαν την γραπτή δήλωση 71-2010 έτσι ώστε να ζητήσουμε ενίσχυση της προστασίας των καρχαριοειδών Πρόκειται για ένα είδος ε, το οποίο ε, κατακρεουργείται στην ε, θάλασσα κυρίως μέσω της αποκοπής των πτερυγίων τους και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που υπερψηφίσατε δηλαδή που υπογράψατε συλλογικά αυτήν την δήλωση ζητώντας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενισχύσει την προστασία του είδους αυτού. Ευχαριστώ Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Περνάμε τώρα στις ψηφοφορίες. Ε,